E, Συνεχίζεται η συνεδρία κύριε και κύριοι. Ο κύριο Πόσελτ, κύριε Πρόεδρε, είστε ένα πραγματικά εξαίρετο πρόεδρο του σώματο, ωστόσο επιθυμώ να διαμαρτυρηθώ για τον τρόπο σχεδιασμού των κοινοβουλευτικών εργασιών από την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζουν ότι σήμερα έχουν λίγα πράγματα στην ημερήσια διάταξη. Γιατί δεν δείχνουν κάποια ευκαμψία να μας δώσουν ε, περισσότερο χρόνο αγορεύσεως. Έχουμε εδώ ε, ανθρώπους όπως τον κύριο Μπρόκ, τον κύριο Σούριαν. Θα ήθελα πολύ να τους δοθεί περισσότερος χρόνος. Πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να μιλήσουν σήμερα εάν, εν πάση περιπτώσει, είχε υπάρξει δυνατότητα να δράσει ο σχεδιασμός του Κοινοβουλίου πιο εύκαμπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσελτ. Θα καταγράψω αυτά που λέτε και θα λάβω υπόψη πολύ σοβαρά την πρότασή σας. Ο αντιπρόεδρος κ. Ρούτσεκ είναι εδώ παρόν, ο οποίος σε δύο λεπτά θα αναλάβει την ε, προεδρία της συνεδρίασης και είμαι σίγουρο ότι θα δώσει άπλετο χρόνο ομιλίας στους ε, βουλευτές εφόσον το έχουν ανάγκη. Ίσως δεν θα μπορέσει να μετατρέψει τα δύο λεπτά σε πέντε, αλλά ίσως θα μπορέσετε να περάσετε κατά 50% τον κανονικό χρόνο μιλία σας. Αντί για δύο λεπτά θα έχετε τρία. αλλά πολλές φορές ακόμα και για δύο λεπτά είναι υπερβολικά τα τρία λεπτά. Μέσα στα πρώτα δύο λεπτά υπάρχει τέτοια ακρίβεια στο λόγο που δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα περισσότερο. Και αν μπορώ να ξεκινήσω, παρακαλώ.